Συνάδελφοι, καθίστε παρακαλώ. Cominciamo a prendere posto. Καθίστε παρακαλώ. Allora, direi di cominciare. Νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε. Καθίστε παρακαλώ. Επαναλαμβάνεται η συνεδρίαση. Στην ημερήσια διάταξη έχουμε την εκλογή του Πρόεδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όπως γνωρίζετε, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρότεινε ως υποψήφια την κυρία Ούρσουλα Φόρντεν Λάιερ για πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Να σας υπενθυμίσω ότι βάρθηση του άρθρου 124 παράγραφος 2 του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σύμφωνα και με το άρθρο 17 παράγραφος 7 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκλέγει τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με πλειοψηφία των μελών που το αποτελούν. Η ψηφοφορία είναι μυστική. Οι οδηγίε για την εκλογή του Πρόεδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχουν διανεμηθεί σε όλους τους ευρωβουλευτές. Χρειαζόμαστε 8 ψηφολέκτε για τη διαδικασία της ψηφοφορίας και από εκεί και πέρα ε, πρέπει να γίνει η κλήρωση. David Ivan. David Ivan. Πού είστε? David Ivan. Δέχεστε? Πολύ ωραία.